Dear colleagues, we can start... Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομική Βοήθεια. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βάλτερ Ράντερμάχερ, που είναι Γενικός Διευθυντής της Eurostat. Ξέρω ότι θα συνταξιδοτηθείτε ε, σύντομα θα ήθελα και εκ μέρου των μελών της Επιτροπής να σας εκφράσω την ε, εκτίμηση και ικανοποίησή μας για τις υπηρεσίες σας ως Γενικού Διευθυντή τη Eurostat και να σας ευχαριστήσω για την ε, θαυμάσια συνεργασία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολύ μεγάλα στατιστικά ζητήματα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις μελλοντικές σα ε, δραστηριότητε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε βεβαίω. Και θα έχουμε μια βιντεοδιάσκεψη. Ε, θα συνδεθούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και θα μιλήσουμε τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου, που ήταν πρόεδρος, όπως ξέρετε, της ε, Ελστάτ από το 2010 μέχρι το 2015. Καλώς ήρθατε κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, γιατί είναι πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεστε. Η συνάντηση αυτή θα έχει ως κεντρικό της θέμα τις ε, στατιστικές, τη σημασία των καλών στατιστικών για την καλή διακυβέρνηση, αλλά και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα το δικό μας, τα προγράμματα δηλαδή οικονομικής βοήθειας. Γιατί για αυτά ασχολούμαστε εδώ και κυρίως ε, για το θέμα της Ελλάδας. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Ραντεμάχια και συνεχεία στον κύριο Γεωργίου για 7 λεφτά ο καθένα για να κάνουν τι εγωγικέ του παρατηρήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επίτροπης, καλησπέρα σας. Με προσκαλέσατε σήμερα εδώ να έρθω ενώπιον της Ομάδας Εργασίας Οικονομικής Βοήθειας για να συνεισφέρω στη συζήτηση όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση για τις επίσημες στατιστικές στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες για την εισαγωγή και την εφαρμογή ε, νέων μέτρων από το 2010. Υπήρχαν προβλήματα ποιότητας με τις επίσημες στατιστικές στην Ελλάδα που πάντοτε αποτελούσαν ε, αιτία ανησυχίας και γι' αυτό ε, πολλές φορές με πρωτοβουλίε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πριν από αυτό το έτος υπήρξαν προσπάθειες ε, αναμόρφωσης του συστήματος. Το 2009 η Eurostat έπρεπε να γύρει μια επιφύλαξη όσον αφορά τον τρόπο που οι ελληνικές αρχές είχαν υπολογίσει το ε, εθνικό έλλειμμα και, την, ε, και το χρέος ε, και τα στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δοθεί σε εμά με την κοινοποίηση για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος τον Οκτώβρη. Στις 2 και 21 Οκτωβρίου η Eurostat έλαβε δύο διαφορετικές ε, πίνακε πίνακες δηλαδή που κάλυπταν τα έτη 2005-2008 και μια πρόβλεψη για το 9. Στην ε, κοινοποίηση του Οκτωβρίου, ε, της 21ης Οκτωβρίου, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, είχαμε αναθεώρηση του ελλείμματος από μείον 5% του ΑΕΠ στο 7,7% του ΑΕΠ. Οι ελληνικές αρχές επίσης αναθεώρησαν την πρόβλεψη ε, για το 2009 από 3,7% του ΑΕΠ όπως αναφέρθηκε δηλαδή την άνοιξη του 2009, στο 12,5% του ΑΕΠ. Λόγω διαφόρων παραγόντων, λόγω της οικονομικής κρίσης, ολισθήσεις στον προϋπολογισμό λόγω κλογών και διάφορες αποφάσεις σε επίπεδο λογιστικό. Οι αναθεωρήσεις αυτού του μεγέθους στα εκτιμόμενα ελλείμματα του παρελθόντος είναι εξαιρετικά σπάνιες στα κράτη-μέλη της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όντως στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές φορές. Η Eurostat λοιπόν ξεκίνησε μία ε, έρευνα μεθοδολογική και επισκέφθηκε την Αθήνα. Το προσωπικό μας είχε ε, σκοπό να ελέγξει τους λόγους που υπήρξε αυτή η ασφαλμένη αναφορά των στοιχείων για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και βράθηκαν μια σειρά από αδυναμίες και προβλήματα στο σύστημα αναφοράς ε, των ε, κυβερνητικών οικονομικών που στην ουσία ήταν η καρδιά του προβλήματος. Η έρευνα οδήγησε σε μια χωρίς προηγούμενο και ιδιαίτερα μεγάλη αναθεώρηση των στοιχείων προς τα πάνω ε, βάσει της κοινοποίησης του Απριλίου του, της 22 Απριλίου του 10. Έτσι λοιπόν το έλλειμμα έφτασε στο 13,6% του ΑΕΠ και 115,1% του, του ΑΕΠ ήταν το χρέος. Και το φθινόπωρο του 10 καταλήξαμε στο μείον 15,4% και 126,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της μεθοδολογικής επίσκεψης δημοσιεύτηκαν αναλυτικά στην έκθεση της 8 Ιανουαρίου του 10 της Κομισιόν και όχι μόνο της Eurostat που μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ. Αυτή η έκθεση ρίχνει φως στα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τον τρόπο που συντάσσονται τα στοιχεία στην Ελλάδα. Βρήκαμε στοιχεία για καταχώρηση εσφαλμένων στοιχείων, μη σεβασμό των ε, λογιστικών κανόνων, κακή συνεργασία και μία ε, αμφίσιμη ενδυνάμωση βασικών εθνικών αρχών σημαντικά προβλήματα στον τρόπο που λειτουργεί το εθνικό λογιστικό σύστημα. Όλα αυτά δείχνουν πολύ κακή διακυβέρνηση στο στατιστικό σύστημα της χώρας, μεθοδολογικά λάθη, κακές πηγές και φυσικά και η θελημένη συμπεριφορά. Πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν επιγόντων. Επιγόντως. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν ξεκίνησε μια έντονη δημόσια συζήτηση που συντάραξε τις οικονομικές αγορές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι επενδυτές, οι πολιτικοί παράγοντες ε, αισθάνθηκαν ότι υπήρξε μια μεγάλη, ένα μεγάλο πλήγμα στις εθνικές στατιστικές της Ελλάδος και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και γενικώ μια συζήτηση για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, το οποίο τέθηκε να αμφιβόλο. Και αυτό ήταν το πιο σοβαρό για μας. Η Κομισιόν παρουσίασε τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας ε, ε, στο ΕΚΟΦΗΝ στις 19 Ιανουαρίου του 2010. Βάσει λοιπόν αιτήματος ε, του Συμβουλίου ξεκίνησε μία ένα κοινό σχέδιο δράσης για τις εθνικές στατιστικές της Ελλάδος, το YOSCAP το 2010, που συμπεριέλαμβανε τρεις πυλώνες το πλαίσιο το θεσμικό και της διακυβέρνησης, την ε, στατιστική ικανότητα σε διάφορους τομείς ε, και τις στατιστικές δημοσίων οικονομικών. Ο πρώτος πυλώνας λοιπόν, ε, μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, διαμορφώθηκε και μεταρρυθμίστηκε από τον Έλληνα νομοθέτη και δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα στην Ελλάδα, η ΕΛΣΑΤ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2011 ε, ανέφερε κάθε δράση μέσα στα πλαίσια του Γιοσκάπ και η Eurostat είχε λεπτομέρειες ε, τις οποίες μπορούσε να παραθέτει στο, στην ε, Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου ε, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η Eurostat επίσης έδωσε τεχνική βοήθεια στην Ελστάτ από το 2010 έως σήμερα, δηλαδή 1.100 ημέρες εμπειρογνωμοσύνης και πάνω από 100 αποστολές εμπειρογνωμόνων. Επίσης, αφιέρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ του λειτουργικού προϋπολογισμού της για αυτή τη βοήθεια. Και φυσικά πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό τους εσωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες της Ελστάτ ε, σε άλλους στατιστικούς τομείς όπως και την τεχνική υποστήριξη που προσφέρουν οργανισμοί όπως το ΔΝΤ. Επανερχόμενοι τώρα στην κατάσταση το 2010, οι ελληνικές αρχές ε, έκαναν μια μεγάλη αναθεώρηση της στατιστικής νομοθεσίας της χώρας. Για αυτή τη μεταρρύθμιση ε, χρησιμοποιήθηκε ο αναθεωρημένος ε, κανονισμός των Ευρωπαϊκών Στατιστικών 22309 που το γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής σας που έθεσε τα νέα στάνταρ για το νέο στατιστικό σύστημα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της νομοθεσίας δημιούργησε τη νέα στατιστική αρχή της Ελλάδος, την Ελστάτη, η οποία είναι αρμόδια για το Εθνικό Σύστημα Στατιστικών και είναι και λειτουργικά ανεξάρτητη, διοικητικά και οικονομικά αυτόνομη και δεν υπόκειται σε έλεγχο από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο διοικητικό όργανο. Ο πρόεδρος της Ελστάτ, ο κύριος Γεωργίου, διορίστηκε και να πω σήμερα ότι πρέπει να τιμήσουμε την μεγάλη συνεισφορά που ο κύριος Γεωργίου είχε στην, στον εξυγχρονισμό, τη μεταρρύθμιση και την σωστή διακυβέρνηση βάσει των ευρωπαϊκών στατιστικών κανόνων που εφάρμοσε το νέο στατιστικό σύστημα της Ελλάδας, κάτι που το χρειαζόταν πολύ η χώρα. Τελειώνοντας, ε, δράτω με της ως ε, τελευταία μου παρουσία εδώ στην Επιτροπή σας να σας μιλήσω για τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από αυτό. Καταρχάς δεν πρέπει να μιλάμε ε, για αυτήν ε, ως, για αυτή την εσφαλμένη αναφορά στοιχείων ως την αιτία της οικονομικής κρίσης. Αυτό ήταν απλώς ένα σύμπτωμα σημαντικών λαθών μιας παροχημένης διαδικασίας που χρησιμοποιούσε η Εθνική Διοίκηση για τα στατιστικά της στοιχεία τότε. Δεύτερον, το ευρωπαϊκά και εθνικά στατιστικά συστήματα χρειάζονται ανεξαρτησία, ικανότητες, διαφάνεια και λογοδοσία. Τρίτον, οι νομικές μεταρρυθμίσεις και στρατηγικές εξυγχρονισμού των ε, στατιστικών διοικήσεων θα είναι επιτυχημένες μόνο αν ενσωματώνονται σε ένα ε, υποστηρικτικό και αξιόπιστο πολιτικό περιβάλλον. Η δημόσια και πολιτική συζήτηση ε, θα πρέπει να προωθεί την ακαιρεότητα, ανεξαρτησία και ισχύ των στατιστικών υπηρεσιών και της αναφοράς των στοιχείων. Η στατιστική είναι θέμα εμπιστοσύνης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η εμπιστοσύνη αυτή μπόρεσε να ξαναοικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει σε εθνικό επίπεδο ακόμα ένα κενό που πρέπει να το ξεπεράσουμε. Υπάρχει αυτή η υποψία, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στις στατιστικές αρχές που παραμένει στην Ελλάδα. Τέλος, οι ευρωπαϊκές και εθνικές Στατιστικέ αρχέ πρέπει και θα συνεχίσουν ε, να απολαμβάνουν τη συνεχούς υποστήριξή σας γιατί τη χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γεωργίου. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ μαζί σα και θα ήθελα να θέσω δύο πρωταρχικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι επί πολλά χρόνια οι ευρωπαϊκέ στατιστικέ που παράγονταν στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούσαν το κοινό μα ευρωπαϊκό δίκαιο και κατά εξακολούθηση και, και προθέσεω ήταν εσφαλμένε, υποσκάπτοντα ε, την πολιτική, τι αγορέ και τη δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντα στην ανάδυση της κρίσης. Τα πέντε χρόνια που ήμουν πρόεδρος της ΕΡΤΣΤΑΤ αυτό το, αυτός ο φορέας ουσιαστικά αναδιοργανώθηκε και οι ευρωπαϊκές στατιστικές στην Ελλάδα παράγονταν με βάση το δίκαιο, υποστηρίζοντας λοιπόν τις προσπάθειες για να επιτευχθεί οικονομική σταθερότητα και ευημερία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιες στατιστικές υποστηρίζουν την παρούσα οικονομική βοήθεια που ζήτησε η Ελλάδα και, την, και που της δόθηκε σε ό,τι αφορά επίσης ε, την χρηματοδότηση του προπολογισμού και την απομείωση του χρέους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι πολυάριθμε διώξει και έρευνε εναντίον μου και εναντίον άλλων που συνεχίζονται επί πολλά χρόνια, καθώ και επίμονε πολιτικέ επιθέσει, καθώ και αποσία υποστήριξη από διαδοχικέ ε, κυβερνήσει, δημιούργησαν αντικίνητρα στου στατιστικολόγου στην Ελλάδα για να παράγουν αξιόπιστε στατιστικές. Ως αποτέλεσμα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονό ότι το πρόβλημα τη Ελλάδα με τι ευρωπαϊκές στατιστικές θα επανεμφανιστεί. Η ζημιά που εμφανίστηκε αφορά όχι μόνο τι επίσημες στατιστικέ στην Ελλάδα, αλλά πιο ευρέως αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά θα χρειαστεί χρόνο για να αντιστραφεί η κατάσταση. Όλα αυτά που λέω δεν τα λέω με χαρά. Είμαι Έλληνα, αγαπώ τη χώρα μου. Επέστρεψα στην Ελλάδα για να γίνω επικεφαλής της Ελστάτ, γιατί ήθελα ε, να βοηθήσω την Ελλάδα και γιατί πιστεύω στη χώρα μου. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Πιστεύω ότι η χώρα μου θα προχωρήσει σε, σε στεναρά θεμέλια και με ανανεωμένη δέσμευση σε αξιόπιστες ε, στατιστικέ και με ειλικρινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, μέχρι τα μέσα του 2010, δεν παρακολουθούσε τι στατιστικέ αρχέ που έχουμε στην ε- Ελλάδα, δηλαδή του κώδικα ορθή πρακτική για τι στατιστικέ ε, υπήρχε ε, έλλειψη ανεξαρτησίας από πολιτικούς φορείς, ε, πολιτικές ε, επιρροές και αναμίξεις, ε, έλλειψη αμεροληψίας, έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας και μη ποιοτικέ στατιστικές. Αυτό έχει βαριέ συνέπειε για την παραγωγή επίσημων στατιστικών. Ανάμεσα στον Απρίλιο του 2005 και τον Απρίλιο του 2010, η Eurostat με τι κοινοποίησεις για τη διαδικασία υπερβολικού έλλειμματος εξέφρασε ε, επιφυλάξει σε 6 από τι 11 αυτέ εξαμηνιαίες δημοσίευση. Επίση, η Ελλάδα ε, δέχτηκε 8 μεθοδολογικέ επισκέψει για να αντιμετωπίσει τα, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των ελληνικών στατιστικών, ενώ κανένα άλλο κράτο μέλο δεν έχει λάβει τέτοιε επισκέψει. Ε, τον Ιανουάριο του 2010 με την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Νοέμβριο του 2010 με την έκθεση τη Eurostat εντοπίστηκαν πάνω από 12 μείζωνα προβλήματα, όχι ένα ή δύο, που αφορούσαν εσφαλμένε ευρωπαϊκέ στατιστικέ για την το, ε, επίσημο έλλειμμα, το κρατικό δηλαδή έλλειμμα και χρέος στην περίοδο από τον Απρίλιο του 2005 μέχρι το 2010. Να σας δώσω και άλλε πληροφορίε. Ε, τα μέσα του 2010 ξεκίνησε μια προσπάθεια για να αναδιοργανώσουμε την Ελστάτ. Ε, όλα αυτά, ε, όλη αυτή την προσπάθεια ε, την αντικατοπτρίζουμε στην έκθεση για τη δουλειά της ε, Ελστάτ που σας την έχουμε μοιράσει. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες υπήρξε μια έντονη ανάκτηση ε, της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών της Ελλάδας. Ε, η Ελλάδα κέρδισε την εμπιστοσύνη ε, και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των ε, κρατών μελών και των ε, διεθνών οργανισμών και των αγορών. Η Ελλάδα επέστρεψε στις, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Υπήρξαν δέκα συναπτές εξαμηνιαίες δημοσιεύσεις ε, χωρί επιφυλάξει από τη Eurostat από τον, Απρίλιο, από τον Αύριο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Αυτέ οι στατιστικέ χρησιμοποιήθηκαν από τέσσερι διαφορετικέ κυβερνήσει σαν βάση για να ασκήσουν οικονομική πολιτική και να προβούν σε διεθνή συνεργασία. Ε, και εδώ συμπεριλαμβάνω και τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που δόθηκε στη χώρα ε, με το δανεισμό 300 δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι το 2016 σε τρία διαδοχικά πακέτα διάσωση. Σε αυτό το κόντεξ θα ήθελα να τονίσω ότι τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ που, δόθηκαν, που ζήτησε η Ελλάδα και που δέθηκαν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν τον Αύγουστο του 2015 βασίστηκαν στατιστικέ που παρήγε η Ελστάτ υπό την αιγίδα μου, χρησιμοποιώντα την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ε, κοινοποίηση διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο του Νοεμβρίου του 2010 για να υπολογίσουμε το χρέο και το έλλειμμα του 2009. Το ίδιο ισχύει και για την απομείωση του χρέους που οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ε, του ζητήθηκε να δώσουν στην Ελλάδα μεσοπρόθεσμα και βράχυπρόθεσμα. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα ε, από την ανάκτηση της αξιοπιστίας ε, στις ελληνικές στατιστικές. Παρ' όλα αυτά, αυτέ οι στατιστικέ που είναι τόσο κεντρικέ για το μέλλον τη Ελλάδο ε, έχουν αμφισβητηθεί και για την ακρίβειά του και για τι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή του. Πολύ συγκεκριμένα, ε, ε, έχω υποστεί μια σειρά από διακαστικές διώξει και αστικές αγωγές, οι οποίε μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ποινική δίωξη εναντίον εμού και δύο ανώτερων στελεχών τη Ελστάτ για την αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειμμα του 2009 και την υποτιθέμενη ζημιά στη χώρα 171 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό επιφέρει ποινή ε, κάθερξη. Επίσης, ποινική δίωξη για την ε, υποτιθέμενη παραβάση καθήκοντο ε, που επιφέρει ποινή δύο ε, ετών κάθερξης. Η δίκη μου είναι στις 6 Δεκεμβρίου. Μια νέα δικαστική έρευνα που ξεκίνησε 1η Σεπτεμβρίου του 2016 και επαναλαμβάνει τις κατηγορίες για το έλλειμμα του 2009 και επίσης μιλάει και για συνενοχή της Eurostat και του Δουνουτού. Επίσης, ε, η κατηγορία για την οποία κατεδικάστηκα τον Ιούνιο του 2016 σε 12 μήνες φυλάκιση είναι ε, αυτή της εγκληματικής δυσφήμισης. Αυτό προέκυψε από μια, ένα δημοσίευμα του Ιουλίου του 2014 στο οποίο οι στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ ε, αναφέρθηκε ότι έπρεπε να γίνονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθών Πρακτικών. Αυτό ήταν το δημοκρατικό μου δικαίωμα για να μιλώ ελεύθερα. Και υπάρχει και μια αστική ε, δίκη γι' αυτό. Αυτές οι υποθέσεις λοιπόν και οι έρευνες ε, στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα για, την, ε, για τους σημερινούς θεματοφύλακες των στατιστικών. Χρειαζόμαστε αξιόπιστες στατιστικές, γιατί όλα αυτά έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο. Αυτές οι προκλήσεις υποσκάπτουν τις προσπάθειες της Ελλάδος να επιτύχει οικονομική σταθερότητα και ευημερία. Είναι μια σειρά από περίεργα προηγούμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι επίσημοι στατιστικολόγοι δεν μπορούν να έχουν ακριβείς επίσημες στατιστικές, τις οποίες στηρούν χωρίς να φοβούνται ότι θα τους επιτεθούν, θα τους, επιτεθούν, θα τους δαιμονοποιήσουν και θα τους σύρουν στα δικαστήρια, τότε η ακεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του οικονομικού τη συστήματος τίθεται ένα αμφιβόλο. Το ίδιο ισχύει και για την αξιοπιστία και σταθερότητα του, εθνικού, του διεθνούς οικονομικού συστήματος η προοπτική της φυλάκησής μου θέτει σημαντικά ζητήματα σε μια δημοκρατική κοινωνία για την Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκει. Επίσης, σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουν σε επίπεδο στατιστικών και στατιστικολόγων. Είναι σοβαρές και θα πρέπει να, να επενδύσουμε μεγάλη προσπάθεια για να τις ανατρέψουμε. Ο κύριος Κίρτσος είναι ο πρώτος ομιλητής. Λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Ραντερμάχερ η τωρινή κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει την τάση να καθυστερεί τις πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα της ε, οικονομίας και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζει μια καλύτερη οικονομική κατάσταση από στατιστική άποψη. Ε, είναι η Ελστάτ λοιπόν και η Eurostat σε θέση να υπολογίσει τις καθυστερούμενες οφειλές του ελληνικού κράτους και να κάνει τις σωστές διορθώσεις ε, βάσει στατιστικών στοιχείων. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα στον κύριο Γεωργίου ο οποίος ε, θα αθωθεί πιστεύω, θα δικαιωθεί. Δεν είναι έτσι η κατάσταση στην Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει να τον βάλει στη φυλακή στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Η Ελστάτ, η ανεξάρτητη λοιπόν στατιστική αρχή, είναι μια αρχή την οποία βοηθήσατε κύριε Γεωργίου να αναδιοργανωθεί από το 2010 και ως το 2015. Σήμερα θεωρείται αποτελεσματική και αξιόπιστη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πολιτική διαφωνία που συνεχίζεται σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 και πώς αυτό αυξήθηκε μετά από τις αλλαγές στους στατιστικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους είχε εκτιμηθεί το 2010. Θα μπορούσατε να συνοψίσετε δύο ή τρεις βασικές αλλαγές στους στατιστικούς κανόνες. Πώς αυτοί επιερέασαν τα επίπεδα του ελλείμματος για τον προϋπολογισμό του 2019 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε την συνάντησή μας σε 30 λεπτά. Πρέπει να ομοδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Η κυρία Περβάνς Μπερέσα. Μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Ράντεμάχερ, σας ευχαριστώ για τα συμπράσματα στα οποία προβήκατε από όλα, αυτά, από όλα αυτά τα θέματα. Είπατε ότι για να υπάρχει εμπιστοσύνη στους ε, στατιστικολόγους για τη δουλειά που κάνουν, έχει μεγάλη σημασία. Θεωρείται ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα παρεμβαίνει, ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα εφαρμόζονται, συνεισφέρουν σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που θα ήταν ευνοϊκό, ούτως ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη στις στατιστικές και στους στατιστικολόγους. Και αν όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε. Παραδόξως, επίσης, έχω και μία ερώτηση προς τον κύριο Γεωργίου, που Ε, είναι σε ευθεία συνέχεια από αυτά που ακούσαμε. Ήσασταν υπεύθυνο το 2010 ως το 2015. Αλλά δεν ξεκίνησαν τότε τα προβλήματα με τις στατιστικές. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Χωρίς να το θέλετε κλείσατε το μικρόφωνο σας. Καρδόνς, πρέπει να ανάψεις το μικρόφωνο σου. Ερώτηση προς τον ε, κύριο, κύριο Γεωργίου. Πέρα από την ε, ευθύνη που αναλάβατε ανάμεσα στο 2010 και το 2015, πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν κάποιοι δισταγμοί σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών ήδη από το 2005. Τελικά, Πώς εξελίχθηκαν τα προβλήματα τα οποία μας παρουσιάσατε, δηλαδή σύν το χρόνο πούμε. Πρώτα ο κύριος ε, Ράντερ Μάχερ και συνεχεία ο κύριος Γεωργίου θα απαντήσει. Η πρώτη ερώτηση του κύριου Κίτσου είναι εάν μπορούμε να πούμε κάτι για τα καθυστερούμενα. Φυσικά, ένα από τα διδάγματα που μάθαμε από την ελληνική ιστορία ήταν αυτό. Το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους απλήρωτους λογαριασμούς, ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει πολλές έρευνες, έχουμε ασχοληθεί, έχουμε εγγύψει του προβλήματος για να δούμε πώς τουλάχιστον θεωρητικά θα πρέπει να αναφέρονται τα καθυστερούμενα από την κυβέρνηση που θα πρέπει να καταχωρούνται και επίσης στην πράξη να παρακολουθούμε και να καθαρίζουμε τα, τους λογαριασμούς εκεί όπου αποθηκεύουμε ας πούμε τα τιμολόγια. Εδώ παραπέμπω και στην υπόθεση της Βαλένθια, όπου η Eurostat βρήκε ότι και στη Βαλένθια υπήρχαν καθυστερούμενα και οι πληρωμές δεν έγιναν με σωστό τρόπο και τελικά δώσαμε πρόστιμο στην Ισπανία για αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτό δείχνει ότι παρακολουθούμε το πρόβλημα. Το ξέρουμε και ότι είμαστε σε θέση να μιλήσουμε και για αυτό το πρόβλημα των απλήρωτων λογαριασμών. Δεύτερον, για το πολιτικό κλίμα. Έχουμε το την οικονομική πλευρά και τη στατιστική πλευρά και τη σχέση μεταξύ τους. Είναι καλή αυτή η σχέση. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια στην παρακολούθηση των προγραμμάτων ε, οικονομικής βοήθειας, τόσο πιο πολύ προσέχουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Υπάρχει ο κανονισμός 223, ο οποίος δίνει στην Eurostat μια πολύ ισχυρή θέση και ανεξάρτητη παράλληλα θέση. Το 2008 ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Τότε ήταν που ανέλαβα τη Eurostat. Εμείς δηλαδή, οι στατιστικολόγοι, έχουμε πολύ σημαντικότερο ρόλο τώρα. Είμαστε ανθεκτικοί, υπάρχει ένα στεναρό σύστημα το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με εκείνου που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις τελικά, με βάση τα δικά μα σχήματα παλογιστικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργίου. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, καταρχάς, αφήστε με να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Κίρτσου σχετικά με τα αίτια αναθεώρησης του ελλείμματος του 2009 σε σχέση με αυτά που συμπεριλάμβαν η κοινοποίηση του Απριλίου του 2010 και αυτά που αναφέρθηκαν στον, το ε, Νοέμβρη του 2010 στη σχετική κοινοποίηση. Όπως είδε, είπε ήδη ο κύριος Ραντερμάγερ, 13,5% του ΑΕΠ ήταν ε, το Νοέμβρη στην κοινοποίηση, ενώ 15,4% ήταν η αναθεώρηση στην επόμενο στάδιο. 1,8% λοιπόν του ΑΕΠ ήταν διαφορά. Σε τι αντιστοιχούσε? Πριν σας πω πολύ σύντομα κάποια πράγματα, να σας πω ότι δεν υπήρξε άλλαγη στους κανόνες. Οι κανόνες δεν άλλαξαν. Οι κανόνες απλώς εφαρμόστηκαν. Οι κανόνες υφίσταντο 15 χρόνια ήδη. Άρα δεν άλλαξαν οι κανόνες, απλώς εφαρμόστηκαν πλήρως για πρώτη φορά το Νοέμβρη του 2010 με την σχετική κοινοποίηση. Τι ήταν αυτοί οι κανόνες που εφαρμόστηκαν και ποια τα αποτελέσματα. Πρώτον, είχαμε αναθεώρηση των ασφαλιστικών ταμείων, τον λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων που οδήγησε σε 0,79% αύξηση του ελλείμματος και αυτό ε, οφειλόταν σε διάφορους λόγους. Πρώτον, ε, δεν είχαν συμπεριληφθεί τα εφάπαξ ε, των ε, δημοσίων υπαλλήλων που έβγαιναν στη σύνταξη επίσης πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ ήταν λόγω διπλογοεγγραφής στο σύστημα. Αυτό οδήγησε σε 0,79% αύξηση, όπως είπα. Το δεύτερο μεγαλύτερο θέμα ε, που αφορούσε αυτή την αύξηση ήταν η αναταξινόμηση των ΔΕΚΟ και άλλων ε, τέτοιων ε, νοποδοδού που είχαν ήδη αναταξινόμηση είχαν ήδη προκριθεί ως θέμα στο παρελθόν, αλλά δεν είχε γίνει αυτή η άσκηση. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό την άνοιξη του 2010 και τι υπήρχε ως ε, ε, περιεχόμενο στην επιφύλαξη του Απριλίου του 2010 ε, που είχε γύρει η Eurostat. Άρα 23 δέκο, εκ των οποίων οι 17 έπρεπε να είναι στη γενική κυβέρνηση χωρίς αμφισημία σύμφωνα με τον κανονισμό 223. Αυτό οδήγησε σε αύξηση 0,74% του ΑΕΠ. Και υπήρξαν και κάποιες μικρές ε, προσαρμογές, ε, ας πούμε, στον ισολογισμό, δηλαδή τον τρόπο που καταγράφονται τα έσοδα και οι δαπάνες στον προϋπολογισμό. 16% του ΑΕΚ και επίσης ε, οι καθυστερόμενες οφειλές που ανέφερε ο κύριος Ραντεμάχερ ε, δεν υπήρξε μεγάλη παρακολούθηση των ε, οφειλών, των πληρωτέων δηλαδή υποχρεώσεων των Υπουργείων και των, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά τα εντοπίσαμε και μπήκαν ε, στον προπολογισμό σωστά, οπότε υπήρξε μια αύξηση 0,23% του ΑΕΠ. Συνολικά 0,8% η διαφορά. Η μεθοδολογία αυτή είναι ακριβώς η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και σήμερα και χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία 6,5 χρόνια συστηματικά. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημα της κυρίας Μπερές. Ε, σε τι βαθμό ε, εκτείνονται τα προβλήματα, αν κατάλαβα σωστά την ερώτησή σας. Ε, το θέμα είναι πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα και σε αυτό το σημείο λυπάμαι, αλλά απλώς θα σας διαβάσω την έκθεση της Eurostat του Ιανουαρίου του 2010. Λέει, η αξιοπιστία των στατιστικών της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με το χρέος και το έλλειμμα ήταν θέμα προσοχής ε, και παρακολούθησης για πολλά χρόνια. Το 2004 ήδη είχε αναφερθεί ασφαλμένη αναφορά στοιχείων για τα έτη 1997-2003. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, τα προβλήματα συνέχισαν και μετά από αυτό, παρά την πρώτη κρίση των ελληνικών στατιστικών το 2004. Συνέχισαν τα προβλήματα χωρίς να μειωθούν καθόλου. Και μεταξύ 2005 και 2010 σε έξι από τις κοινοποιήσεις η Eurostat έγιρε ε, επιφυλάξεις. Όταν ε, σταμάτησαν οι επιφυλάξεις, ε, αυτό συνέβη μετά, τις, μετά την ε, επέμβαση της Eurostat και τη διόρθωση. Νομίζω ότι όλα αυτά δίνουν μια πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ. Ροπέρτο Λούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση και για τους δύο ομιλητές. Αυτά που διδάχτηκα από αυτά που μας είπατε είναι σε αυτές τις ε, εκατοντάδες αποστολές που έκανε η Eurostat στην Ελλάδα βρέθηκαν πάρα πολλά λάθη. Καταρχάς, την λογιστική μεθοδολογία ε, μερικές φορές λόγω έλλειψης γνώσης, μερικές φορές λόγω έλλειψης επικοινωνίας, έλλειψης συνεργασίας, ε, λόγω δίπλο εγγραφών κτλ. Όλα αυτά τα είπατε. Να, τώρα ε, υπάρχουν ακόμα αυτά τα λάθη. Αν όμως ε, υπήρχε πραγματική ανεξαρτησία, δεν θα έπρεπε. Η ερώτησή μου είναι, έχετε σκεφτεί μήπω υπήρχε πολιτική πρόθεση πίσω από αυτά τα λάθη. Δεν ήταν απλώ τυχαία λάθη τα οποία ε, έγιναν λόγω έλλειψη γνώση ή λόγω έλλειψης συντονισμού. Ίσως υπήρχε πολιτική βούληση που οδήγησε σε αυτά τα λάθη εκ προθέσεως. Αν έχετε μία υποψία ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη, τότε τα νομικά βήματα που θα πρέπει να ληφθούν εναντίον στατιστικολόγων, ε, εναντίον του κ. Γεωργίου, ο εκφοβισμός που ασκείται, ε, ίσως δηλώνουν ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση πίσω από αυτά όλα αυτές τις κινήσεις. Πιστεύει, πιστεύετε ότι οι τρεις πυλώνες που αναφέρετε επαρκούν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, αρκεί να έχουμε καλύτερη αναγραφή, ε, καλύτερους κανόνες ή μήπως η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική βούληση των παλιών ε, πολιτικών και ηγετών της Ελλάδας ή και των σημερινών. Ο κύριος Αχτουή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Γιατί καταδεικνύει κάποιες ελλείψεις για τον τρόπο διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Καταρχά, να σας πω κύριο, κύριε Ανδρέα Γεωργίου, ότι σα έχω συναντήσει φυσικά το Φεβρουάριο του 2012. Ο Γάλλος πρωθυπουργό το, ο τότε, μου είχε πει να ασχοληθώ ε, με το μέλλον της Ευρωζώνης και άρα να επισκεφτώ διάφορε ε, χώρες της Ευρωζώνης. Ε, Είχα δει τότε, εσά κύριε Γεωργίου, ε, με μεγάλη μου θλίψη είχα δει την κατάσταση στην οποία βρισκόσασταν, γιατί είχατε πει την αλήθεια και όμως αυτό σας, θα σας καταδίκαζε. Κύριε Γεωργίου, είμαστε στο πλευρό σα. Πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια στους δημόσιους λογαριασμούς, στις δημόσιες στατιστικές και θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή ασυλίας των αρχών και υπευθύνων για τις στατιστικές, ούτως ώστε οι πολιτικοί σε καμία περίπτωση να μην προσπαθούν να επηρεάζουν τις στατιστικές τους κατά τη δημοσίευση των δεδομένων. Κύριε Γεωργίου, υπήρξε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά από το 2012 και μετά. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Στατιστικές ε, του 2009-2023 γίνεται πιο σεβαστός. Ε, δεν έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ψηφίζουμε γρήγορα γρήγορα στην Ελλάδα τους νόμους για να είμαστε σύμμορφοι, αλλά δεν εφαρμόζονται τελικά αυτό οι νόμοι και ελπίζω να μην ε, θυμώσουν μαζί μου οι Έλληνες συνάδελφοι. Τέλος, κύριε Γενική Διευθυντά της Eurostat, θα σας ρωτήσω το εξή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση των δεδομένων για τα δημόσια λογιστικά. Γιατί στη Eurostat έχουμε λίγους ε, εμπειρογνώμονε για τα δημόσια ε, λογιστικά, αλλά έχουμε πάρα πολλούς εμπειρογνώμονε και στατιστικολόγου για τα μακροοικονομικά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός τη αρχής των δημοσίων λογιστικών, ούτω ώστε να υπάρχει μια αξιόπιστη εικόνα των δημοσίων λογαριασμών στις χώρες της Ευρωζώνης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη, απόλυτη ανεξαρτησία σε, σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τους δημόσιους λογαριασμούς για να μπορούν να δημοσιεύουν τα δεδομένα τόσο ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισημία. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να είναι ο τόπος όπου θα μπορούσαμε να σχολιάζουμε αυτούς τους δημόσιους λογαριασμούς και ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζονται. Ευχαριστώ. Παρακαλώ συνάδελφοι, και εσείς αγαπητοί φιλοξενούμενοι, να είσαστε πιο σύντομοι. Θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε τι ερωτήσει, γιατί σε 13 λεπτά πρέπει να κλείσουμε τη συνάντηση. Ο κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή όσα είπε ο κύριος Ράντερ Μάχερ και ο κύριος Γεωργίου και τους ευχαριστώ. Θα θέλω να πω ότι τα μαγειρέματα των ελληνικών δημόσιων στατιστικών ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η ελληνική κυβέρνηση σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της Ελστάτ και εγγυάται σε πλήρη και άριστη συνεργασία και με την Κομισιόν και με την Eurostat την ακρίβεια των δημόσιων στατιστικών και είναι δεσμευμένη και προσιλωμένη στην εφαρμογή του προγράμματος με βάση αυτές τις δημόσιες στατιστικές για την ταχύτερη ολοκλήρωση του προγράμματος και ιδιωκότερα της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό δεν είναι δική μου δήλωση. Είναι δήλωση του αρμόδιου Υπουργού κυρίου Χουλιαράκη πριν λίγες εβδομάδες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σημειώσατε και οι δυο σας ότι αυτά τα πολύ δυσάρεστα μαγειρέματα των δημόσιων στατιστικών αφορούν μια περίοδο του παρελθόντος και πρέπει να μείνουν εκεί. Προσθέτω επίσης ότι αυτή η κυβέρνηση ενίσχυσε την ανεξαρτησία της Ελστάτ με νόμο που ψήφισε το καλοκαίρι του 2015 και ότι επίσης το compliance report της Κομισιόν τον Ιούνιο του 2016 καταγράφεται η ενίσχυση της συνεργασίας για την αξιοπιστία των δημόσιων στατιστικών. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Ράντερ Μάχερ είναι πώς αξιολογείται, κύριε Ράντερ Μάχερ, το σημερινό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στην Eurostat και την Ελστάτ για την παραγωγή των σημερινών δημόσιων στατιστικών. Και επίσης τον κύριο Γεωργίου, πώς αξιολογείται τη δουλειά της σημερινής διοίκησης της Ελστάτ που σας διαδέχθηκε πριν λίγο καιρό. Και να προσθέσω για τους συναδέλφους ότι πριν λίγες ημέρες ο αρμόδιος εισαγγελέα κατέθεσε απαλλακτική πρόταση ε, υπέρ του κυρίου Γεωργίου για τις κατηγορίες που κατατέθηκαν στο παρελθόν εναντίον του. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, ο κύριος Βαν Σβέν Καταρχάς, ε, να πω ότι το να ακούμε την ιστορία που μας διηγείστε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κανονικά, οι στατιστικολόγοι πρέπει να προστατεύονται από τις διώξεις. Αυτό ε, είναι εγγεγραμμένο στο νόμο, στο νομικό σύστημα και μας ανισχύει ιδιαίτερα. Πέρα από αυτό, έχω μια ερώτηση και για τους δυο σας. Πώς κρίνετε την τρέχουσα κατάσταση των ε, ελληνικών στατιστικών. Ο συνάδελφος, ο κύριος Παπαδημούλης, ήδη ρώτησε πώς τη βλέπετε, αλλά θέλω να ακούσω την κρίση σας. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση, η ποιότητα του συστήματος. Ήμουν σκιώδης όταν εγώ και κάποια άλλη εδώ στην αίθουσα ψηφίσαμε ε, την έκθεση για την μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών στατιστικών μέσα στα πλαίσια του εξαπτύχου. Και στην ιστοσελίδα της Eurostat Αναρωτιέμαι τώρα αν θα πρέπει να έχω εμπιστοσύνη σε κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα και όπως ε, είπατε και εσείς κύριε Ράντερ Μάχερ, θα ήθελα να μάθω ποια είναι αυτά. Όταν έχουμε εταιρείε με δημόσιες εταιρείε με παθητικό, Έχουμε ας πούμε κάποιες εταιρείες οι οποίες στη Γερμανία, στην ε, Γαλλία δεν μας δίνουν τρέχοντα στοιχεία. Ε, δεν μας δίνουν στοιχεία παρά μόνο μέχρι το 2013. Το ίδιο γίνεται και με την Κύπρο. Επίσης για τις μη ε, χρηματοπιστωτικές εταιρείες ε, και άλλες, τις άλλες εταιρείες που έχουν ζημιές υπάρχουν προβλήματα. Στη Γερμανία, επίσης στη Βουλγαρία, Δανία, Λιθουανία, Φιλανδία, πολλές χώρες μην με διακόπτετε, τελειώνω. Δεν δίνουν καθόλου στοιχεία. Όταν έχουμε λοιπόν αυτή την έμεση μορφή, όχι την άμεση απόκρυψη στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα, ε, νομίζω ότι τα στοιχεία της Eurostat δεν έχουν συνέπεια και δεν έχουν και την κατάλληλη ποιότητα. Πότε θα έχουμε λοιπόν μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ποιότητας των στοιχείων. Ευχαριστώ κυρία Εύα Καϊλή. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου για την παρουσία σας εδώ. Η περίπτωσή σας είναι απόδειξη ότι στην Ελλάδα ένα από τα προβλήματα πάντοτε ήταν η συνεχής προσπάθεια των κυβερνήσεων να χειριστούν και να χειραγωγήσουν τις αρχές. Στο παρελθόν όντως δεν υπήρχε σεβασμός. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ασκήσει πίεση τώρα και να αφαιρέσει αρμοδιότητες από τις ανεξάρτητες αρχές, από τη δικαιοσύνη. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, πάλι θεωρίες συνωμοσία για να αποφευθούν οι ευθύνε, χάνουμε την αξιοπιστία μας συνεχίζοντας αυτή τη θεωρία και κρύβοντας αυτά που συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ε, Θεωρείτε ότι θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο να υπάρξει συμφωνία και να διαπραγματευτούμε ε, το νέο ε, μνημόνιο. Ευχαριστώ. Ο Φάμπιο Ντεμάση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ακριβείς και ανεξάρτητες στατιστικές είναι το κλειδί για να μπορεί κανείς να ενημερωμένος πλέον να λαμβάνει σωστές πολιτικές αποφάσεις. Ε, και εσείς κύριε Γεωργίου αυτό συνεισφέρατε σύμφωνα με την αναφορά της ε, διαδικασίας υπερβολικού ε, για το 2010 στη σελίδα 15 στο, ευρωπαϊκό, στο ελληνικό έλλειμμα ε, συμπεριλήφθηκαν στοιχεία μετά από την ε, επέμβαση της Eurostat που δόθηκαν από την Goldman Sachs. Γιατί αυτά δεν είχαν συμπεριληφθεί πριν και τι έχει γίνει σε άλλες χώρες αντίστοιχα μετά από αυτό. Δεύτερον, υπήρξε μια διαδικασία τον Οκτώβριο του 2010 που ε, προσπάθησαμε να καταγράψουμε την, ε, το κατά πόσο ήταν ολοκληρωμένα τα στοιχεία των ΔΕΚΟ, ε, δηλαδή αν υπήρχε έλλειμμα ή πλεόνασμα. Το 2009 το πλεόνασμα για τις ΔΕΚΟ αρχικά, αρχικά ήταν 125 εκατομμύρια, αλλά τα επόμενα έτη αναθεωρήθηκε το νούμερο και φτάσαμε στα 201 εκατομμύρια, δηλαδή μεγάλη διαφορά. Μπορείτε να μας πείτε γιατί ήταν απαραίτητες αυτές οι αναθεωρήσεις ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ που ενεπλάκησε αυτό, ε, ποιες ήταν οι αιτιολογίες και γιατί κάποιες ΔΕΚΟ προσέβαλαν τις αποφάσεις ε, του κυρίου Γεωργίου ε, για να μπουν στη γενική κυβέρνηση διάφορα πράγματα όπως το Μέγαρο Μουσικής κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το λόγο τώρα στους ε, ομιλητές μας. Πρώτος ο κύριος Γεωργίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με την τεχνική ερώτηση του, του κύριου Ντεμάτζιο. Σε ό,τι αφορά τις off-market swap, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια κατευθυντήρια γραμμή από τη Eurostat την άνοιξη του 2008 για το πώς να χειριστούμε τα off-market swap στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από εκτενείς συζητήσεις που είχαμε στους, ε, στην ομάδα εργασίας ε, για τους οικονομικούς λογαριασμούς όπου συμμετείχε η Ελλάδα. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτά τα swaps, δηλαδή swaps που έχουν ε, τιμή στην αρχή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, να συμπεριληφθούν ως μορφή του χρέους. Η Eurostat και όλες οι χώρες της Ένωσης συμφώνησαν. Υπήρχαν διάφορες χώρες που είχαν τέτοια off-market swaps. Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, μεταξύ άλλων. Και δηλώνουν τα swaps, τα δήλωσαν και τροποποίησαν τους λογαριασμού τους. Αυτό είναι δημόσια. Δημόσιες πληροφορίες. Τότε η Ελλάδα είπε ότι δεν είχε, αλλά είχε στην πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο ήταν το swap της Goldman Sachs. Είπε ότι δεν είχε κανένα και μετά αυτό το θέμα ανέκυψε ξανά μετά από πληροφορίες που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις αρχές του 2010. Ε, εκφράστηκε επιφύλαξη τον Απρίλιο του 2010 στην κοινοποίηση για τη δικασία υπερβολικού έγκληματος από τη Eurostat για τα ελληνικά στοιχεία. Και εγώ όταν ανέλαβα στην Ελλάδα την ηγεσία της Ελστάτ, τότε ε, δέχτηκα να, να, να αλλάξω τα στοιχεία ε, με βάση τους κανόνες που ισχύαν από το 2008 και τα λοιπά και μετά. Αυτό έπρεπε να κάνουμε, τίποτα δεν θα έπρεπε να γίνει διαφορετικό για την Ελλάδα από ό,τι για άλλες χώρες. Η Ελλάδα έκανε ότι έπρεπε να κάνουν και άλλες χώρες. Αυτό ε, προσέθεσε 5,5 δις στους υπολογισμούς του κρατικού χρέους και αυτό γίνεται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Για το θέμα που αναφέρατε, αν το κατάλαβα καλά, μιλάτε σε μια αλλαγή που έγινε, κύριε Ντεμάτζιο, για τις ΔΕΚΟ. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και οι συκοφάντες μας το χρησιμοποιούν για να κάνουν επικρίσεις. Είναι ανακατανομή ε, και περνάνε στον προπολογισμό του, του, της Γενικής Κυβέρνησης. δεν έχει επιπτώσει καθόλου στο έλλειμμα αυτό. Αυτή η ανακατανομή την οποία κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο τεχνικό σας θέμα, δηλαδή πώς υπάρχουν φορείς που πήγαν στο διοικητικό δικαστήριο για να αμφισβητήσουν την ε, ταξινόμησή τους, αυτοί οι φορείς υπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια πολλοί από αυτούς. Όταν το πρόγραμμα προσαρμογής όμως άρχισε να τρέχει, υπήρχαν περιορισμοί. Και αυτοί οι φορείς δεν, θεώρησαν ότι είναι θετικό να μπουν στο γενικό προπολογισμό. Και γι' αυτό πήγαν στο διοικητικό δικαστήριο. Τα κριτήρια για συμπερίληψη αυτών των φορέων στο γενικό προπολογισμό τη κυβέρνηση έγινε μετά από την, από την επανεξέταση που έκανε η Eurostat μετά από πολλούς μήνες και η Elstat χρησιμοποίησε τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούν ε, και οι υπόλοιπε ε, στατιστικές υπηρεσίες στις άλλες χώρες. Αυτό το συγκεκριμένο τεχνικό θέμα, αυτή η τεχνική προσέγγιση, ε, σε 13 διαφορετικές κοινοποίησεις ε, εξετάστηκε από την ε, Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Τώρα, για το αν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, για το αν άλλαξαν τα πράγματα. Ο κύριος Ζαντερμάχε είπε κάτι πολύ σημαντικό νομίζω, ότι το θέμα δεν είναι τι κάνουν μόνο οι στατιστικολόγοι, είναι και το πολιτικό περιβάλλον και πώς λειτουργεί. Και πώς λειτουργούν οι στατιστικολόγοι μέσα στο πολιτικό κλίμα. Και κατά πόσον ο πολιτικός κόσμος υποστηρίζει τους στατιστικολόγους και τη δουλειά του. Ε, μοίρασα ή μάλλον ζήτησα από το γραφείο του Προέδρου να μοιράσει α, αυτό το κείμενο. Τις δεσμεύσεις τι στατιστικές. Το Φεβρουάριο του 2009 το είχε υπογράψει ο Έλληνα Πρωθυπουργό και ο τότε ε, Ευρωπαίος Επίτροπος Υπεύθυνος για τι. Στατιστικές. Και λέει τα εξή ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται επίσημα να εγγυηθεί την επαγγελματική ανεξαρτησία του ελληνικού συστήματος στατιστικών και της Ελστάτ και να προωθήσει μέσω κατάλληλων κοινοποίησεων κάτι τέτοιο. Να υποστηρίξει την Ελστάτ ε, ούτω ώστε να ανακτηθεί η δημόσια εμπιστοσύνη σε ελληνικέ στατιστικέ και να ε, την υπερασπιστεί απέναντι στι προσπάθειε που γίνονται για να υποσκαθεί η αξιοπιστία τη. Επίσημη δέσμευση. Τώρα, αν έχουν γίνει σεβαστέ αυτέ οι δεσμεύσει, Υπάρχει ο 1451 του 2012 στην Ελλάδα που υποτίθεται ότι ακολούθησε αυτή τη δέσμευση, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει σεβασμός αυτής της αρχέ. Στην ε, παρουσίασή μου σας μίλησα για τις διάφορες διώξεις ε, που έχω υποστεί και κάποιοι άλλοι συναδελφοί μου, επειδή ακριβώς κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Υπάρχει μια, ένα όργιο επιθέσεων ενάντια στους στατιστικολόγους και υπ' αυτή την έννοια εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικοί κινδύνοι για τις ελληνικές στατιστικές αλλά και για όλους τους στατιστικολόγους ανά τον κόσμο. one Ωραία. Να επανέλθω λοιπόν στις δύο ομάδες ε, ερωτήσεων. Το παρελθόν και το παρόν. Η κατάσταση του 2009-10 εάν είναι συγκρίσιμη με τη σημερινή. Και θα έλεγα όχι. Σε καμία περίπτωση δεν έχω αυτή την άποψη. Η κατάσταση τώρα δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή που είχαμε το 2009. Όταν μιλάμε για αδυναμίες στο ελληνικό στατιστικό σύστημα σήμερα, είναι τεχνικές αδυναμίες, ε, ε, αδυναμίες εφαρμογής, αδυναμίες σε επίπεδο ικανοτήτων, δεξιοτήτων, τέτοια πράγματα. Δεν είναι αυτό που βρήκαμε το 2009, δηλαδή η θελημένη ε, αναφορά εσφαλμένων στοιχείων. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα λοιπόν αν μπορούσαμε να κλείσουμε τα πάντα συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων του, εναντίον του κυρίου Γεωργίου, να τα βάλουμε στο παρελθόν. Περασμένα, ξεχασμένα, κοιτάμε τώρα την κατάσταση που έχουμε το πολιτικό περιβάλλον στην Ελστάτ, που περιβάλλει την Ελστάτ, να δώσουμε στην Ελστάτ την ικανότητα ε, τις δεξιότητες, την πρόσβαση στα στοιχεία, τα διοικητικά, τα, η οποία θα μπορέσει να την βοηθήσει να υπερβεί τα εμπόδια όπως γίνεται και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα έπρεπε να γίνει επίσης μια εκστρατεία επιτόπου, ένα μάρκετινγκ που θα δι θα διαφημίσει ας πούμε την Ελστάτ στους Έλληνες πολίτες. Θα τους πει ότι πρέπει να την εμπιστεύονται πλέον. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι κάτι που ε, εύκολα χάνεται αλλά δύσκολα ανακτάται. Αυτό είναι που πρέπει να ανακτήσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει στη χώρα. Με χαρά μας όμως θα βοηθήσουμε. Τώρα, Δεύτερον, τι μπορούμε ως στατιστικολόγοι να κάνουμε για να εγγυηθούμε ότι και για τα μικροστοιχεία δεν υπάρχουν σφάλματα. Αυτά τα είπε και ο κύριος Γκίγκολτ και άλλοι συναδελφοί σας. Εμείς στην Eurostat έχουμε 850 άτομα στο προσωπικό μας. Ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εθνικές στατιστικές αρχές ε, συνολικά έχουν 50.000 άτομα η Eurostat δεν μπορεί να αντικαταστήσει ε, τους ε, επιτόπου ελεγκτές, να είμαστε οι ελεγκτές των ελεγκτών. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε ένα Λουξεμβούργο. Είμαστε ένα σύστημα στατιστικής με διάφορα επίπεδα. Και αυτό ε, περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τη στατιστική νομοθεσία που πέρασε πριν από δύο χρόνια. Επίσης υπάρχει ένα project, το λεγόμενο EPSAS, το οποίο προσπάθησε να προχωρήσει και να μπει στο θέμα των δημόσιων οικονομικών σε μικροεπίπεδο, δηλαδή σε κάθε δήμο, σε κάθε νησί, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Ο κάθε δήμαρχος πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα δημοσίων, δημοσίας, ε, λογιστικής, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία, να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και σε μικρότερη κλίμακα, όχι μόνο δηλαδή στους εθνικούς λογαριασμούς. Στο μικρότερο αυτό επίπεδο λοιπόν που ανέφερε ο κύριος Γκίκολτ, ε, δεν έχω χρόνο να επανέλθω στην ερώτησή σας, αλλά με χαρά μου δεσμεύομαι εγώ και το, το όργανο που εκπροσωπώ να συντάξει μια έκθεση για το θέμα που έθεσε ο κύριος Γκίκολτ. Ε, όχι ακριβώ έκθεση, λέει ο κύριος Κίκολτ, απλώς να απαντήσετε γραπτώς στο ερώτημα. Τι έγινε με τα επιπλέον στοιχεία της έκθεσης Φάουλ. Και μια χαρά θα είναι αυτό για μας. Πρώτα θα κατανοήσω καλά την ερώτησή σας και μετά θα σας δώσω μια πλήρη απάντηση, λέει ο κύριος Ράντερ Μάχερ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράντερ Μάχερ και κύριε Γεωργίου ήταν πολύ χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και σημαντική η ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι πραγματικά αναδύεται και η ξεκάθαρη υποστήριξη αυτής της ομάδας εργασίας ε, ως προς την ανεξαρτησία και την ποιότητα των στατιστικών και των στατιστικολόγων. Επίσης, ένα καλό στοιχείο είναι το τελευταίο σχόλιο του κυρίου Ραντερμάχερ ότι η κατάσταση τώρα δεν έχει καμία σύγκριση με το παρελθόν. Θα ήθελα να συνταχθώ σε αυτό που είπε και να πω ότι πρέπει να κλείσει το παρελθόν. Όλα τα στοιχεία, όλα τα πράγματα που μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα, όχι μόνο τον Σβέν αλλά όλους μας. Κλείνουμε το παρελθόν και με βάση το νέο κανονισμό που εμείς μαζί φτιάξαμε και εγκρίναμε έχουμε εισαγάγει νέα στοιχεία και δουλεύουμε επιτόπου και στην Ελλάδα αλλά και παντού για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλές και αξιόπιστες στατιστικές ως βάση για την καλή και ποιοτική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον κύριο Γεωργίου για άλλη μια φορά και για άλλη μια φορά να τιμήσουμε τον κύριο Ράντερ Μάχερ και να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά του. Αφού απαντήσατε λοιπόν και στην ερώτηση του κύριου Κίκολ, το περιμένουμε να σας ξαναδούμε. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 6 Δεκεμβρίου στις 12.30 με τον κύριο Χουλιαράκη. Πέρα στη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργίου για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ και εγώ.